Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δώσε ένα χρονικό περιθώριο, λόγω και των απεργιών σήμερα, αλλά μια και βλέπουμε αρκετούς συναδέλφους εδώ και προσωπικά βεβαίω. Εμείς οι βουλευτέ μπορεί να μένουμε και πιο κοντά και να έρθουμε με τα πόδια. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σημείο 1, ενεά Αντιμετώπιση τη νομοποίησης παράνομων εσόδων. Ε, ποινικό δίκαιο. Δεν είναι εδώ εισηγητής, άρα πάμε στις ψηφοφορίες μας. Δεν ψηφίζουμε την τροπολογία Τέσσερα. Α, Ιγνάσιο. Καλώς το να. Λοιπόν, κάθισε, όσο να καθίσει εγώ θα κάνω τη δοκιμή των ε, ηλεκτρονικών συστημάτων μας για την ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Α, δεν δουλεύει. Καλά δουλεύει. η ψηφοφορία. Πέρας. Εντάξει, δουλεύει. Έτσι άφησα και το χρονικό περιθώριο στον Ινιάσιο. Το 9. πολέμηση της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. έχει να πεις κάτι. Όχι μόνο ευχαριστώ τους και όδης για τη συνεργασία. Ωραία σύντομα και απλά. Είναι και μεγάλες ψηφοφορίες σήμερα. Υπαριθμών 5 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 5. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθη. 38 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά στο δούμε 38 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε λοιπόν. Άλλες ήταν οι πλειοψηφίες. Η 7 έχει αποσυρθεί. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατάλαβα. Δεν βλέπετε εσείς το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στις δικές σας οθόνες. Παρακαλώ το τεχνικό να μας δείξει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών στις οθόνες. 12 ε, υπέρ, 13 κατά. Η τροπολογία υπαριθμών 10 υπέρ, κατά. Άποχες. Για να επαληθεύσουμε τη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και απερίφθη. 12 υπέρ, 13 κατά. Εξακολουθείτε να μην βλέπετε τα αποτελέσματα. Συμβαστική παριθμών 1 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ, α, ε, κάποιος έχει πάει στο τεχνικό, εντάξει. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ κατά. Αποχές και επαληθεύουμε την 1 παρακαλώ γιατί μάλλον απορρίπτεται από ό,τι βλέπω. Δεν φαίνεται να ήταν τόσο συμβαστική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. 14 υπέρ, 11 κατά. Α, τώρα βλέπετε τα αποτελέσματα της οθόνες, ωραία. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά. Αποχές επαληθεύουμε. 42, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Και εγκρίνεται. Παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά επαληθεύουμε συμβαστική 3 μάλλον έχει εγκριθεί αλλά για να δούμε Πέρασε. πέρασε λοιπόν 13 υπέρ 11 κατά 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε τη 19 παρακαλώ άρχεται 13 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε παρακαλώ την 22. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 13 υπέρ, ε, κατά 12 υπέρ. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές επαληθεύουμε την 26. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη 28 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29η υπέρ κατά. Αποχές, ε, πάλι θεύμα παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, για να επαληθεύσουμε την 30 υπέρ. Ε, άρχεται ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας. Και απερίφθη με διαφορά. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά κατευθείαν. Πέρας και εγκρίνεται. Παρακαλώ τουλάχιστον να βλέπω τι, προς ποια κατεύθυνση ψηφίζουν οι ομάδες, πράσινοι, γκουε. Θα ήθελα ή μη τι άλλο, αν είναι αποχή φερρυπή, να βλέπω καθαρά τη στάση της ομάδας. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την συμβαστική 7 ψηφίσατε όλοι και πέρασε και έχει απορριφθεί ε, η τρια υπέρ κατά αποχές ε, επαληθεύουμε την 3 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορια Απερίφθη. Ίσα ίσα. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 34 γιατί είναι μια μικρή ομάδα που δεν βλέπω πώς ψηφίζει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εύκολο αυτό. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το επαληθεύσουμε παρακαλώ στη συμβαστική 9. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ωραία, εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ίσα ίσα. Μάλιστα. Απερίφθη δηλαδή. Δύσκολο. Δεν προλάβατε εσείς, αλλά είχα πει ότι τέλειωσε η ψηφοφορία. Δεν προλάβατε. Πρέπει να προσέχετε, συνάδελφοι. Οι άλλες ομάδες, αν συμφωνούν να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, το δέχεστε. Καλώ, συνάδελφοι, εντάξει. Στην ε, Ολομέλεια να ξέρετε ότι δεν συμβαίνουν αυτά, βέβαια. Λοιπόν, γίνεται πάλι ονομαστικά η τελική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Παρακαλώ όμω να προσέχετε όλοι. Μερικές φορές βλέπω ότι κάποιος δεν έχει ψηφίσει, αλλά όταν έχω πει δύο φορές ψηφίσατε όλοι, μπορώ να θεωρήσω ότι δεν θέλατε να ψηφίσετε. Και έτσι κλείνονται οι ψηφοφορία. Λοιπόν, όποιο θέλει να ψηφίσει, παρακαλώ, α ψηφίσει. Πέρα τη ψηφοφορία. Και εγκρίνεται με μία ψήφο. Ωραία, τώρα θα πάει και στην άλλη επιτροπή που θα αποφασίσει. Σε ευχαριστώ θερμά και παρακαλώ στην τελική ψηφοφορία ιδιαίτερα να προσέχετε. Ήταν μεγάλη καλοσύνη που δείξατε προ τον εισηγητή μα. Συνάδελφοι, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Πριν όμως θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Θα ψηφίσουμε το 10, Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής Μειώθηση για την Ανάπτυξη. Ο Μωρίς Πόγκα έχει το λόγο που είναι και εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να παρέμβω, διότι παρενέβη χτες ε, και μίλησα και ευχαρίστησα και τους σκιώδεις. Εντάξει, πολύ αποτελεσματικός. Λοιπόν, επειδή θα περνάμε από τη μια σελίδα στην άλλη, τροπολογία 44 να προσέχετε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε την 64 άρχεται η ψηφοφορία.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 εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 97 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, πέρασε. Απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102. Α, απορρίφθηκε. Εντάξει, εντάξει. 102 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 123 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές. Ελέγχουμε τη συμβαστική 22, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και εγκρίνεται. Σας παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι ευκρινώς. 164 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 56, παρακαλώ να δείχνετε τι ψηφίζετε. Δεν ήξερα ότι το ΕΛΚ ε, απορρίπτει. Πέρας, απορρίπτεται έπρεπε να ελέγξουμε. Παρακαλώ όλες οι εβδομάδες να δείχνουν ένας από κάθε εβδομάδα. 168 ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, α, καταπίπτει. 169 υπέρ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά, αποχές, ελέγχουμε την 185, άρχεται η ψηφοφορία, δεν ήταν σαφής οι ενδείξεις από τις ομάδες, απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 194 Α, μόνο το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε. Ωραία, το πρώτο καταπίπτει. Υπέρ του δεύτερου τμήματος, κατά 194 πάντα. Λοιπόν, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σελίδα 19 στο δικό μου κατάλογο, συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε τη 229. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, Α, ξεχωριστή ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Πρώτο τμήμα. Α, καταπίπτει το πρώτο τμήμα, άρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 85. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 40. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 255. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 41. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δυο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ζητούμε μαζί. Αν μπλοκ μπορούμε. Όχι μου λένε. Ωραία. Τρία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία έξι υπέρ, α, καταπίπτει. Ωραία. Επτά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις 8. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές ε, ξανά παρακαλώ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, έκανα λάθος λέει. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε την 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ λοιπόν, παράγραφος 18, την ψηφίζουμε σε τμηματική, πρώτο τμήμα, υπέρ αφετ πια. Πρώτο τμήμα της παραγράφου 18, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ίντα. Γνωμοδότησε της Ίντα. Τα περισσότερα καλύπτονται από τις συμβαστικές. Αιτιολογική α είναι τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. D. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. E. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε. Παράγραφος 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 18 της Λίμπε υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε την έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί για την στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρικής με ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι όσοι επιθυμείτε βεβαίως. Πέρασε. Και εγκρίνεται 19 υπέρ 5 κατά Τρεις αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Πόγκα. Ήταν μεγάλη η πλειοψηφία. Okay, before Πρωτού ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή σε ένα λεπτό, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι ε, μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα σχετικά ε, με την αποδοχή ορισμένων ε, τροπολογιών, διότι πρόκειται για αναδιατύπωση. Όταν πρόκειται για αναδιατύπωση, υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές και όχι μόνο διατύπωσης εκεί όπου υπάρχει μια μικρή αλλαγή μπορεί να μην γίνει παραδεκτή. Εάν ε, η, επιτροπή, βασική επιτροπή το κρίνει, που είναι η Επιτροπή Ήτρε, τότε θα ψηφίσει εκείνη για το θέμα αυτό. Θα αφήσουμε όμως ε, τις αποφάσεις αυτές ε, στην υπεύθυνη, στην αρμόδια Επιτροπή δεν ξέρω, ίσως άλλες επιτροπές να μην κρίνουν το ίδιο όπως θα κρίνουμε κι εμείς. Θα δίνω λοιπόν το λόγο ε, στον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, απλώς να πω ότι σε αυτή τη γνωμοδότηση ήταν δύσκολο να φτάσουμε σε συμβασμούς γιατί είναι ανταγωνιστικές οι θέσεις, αντιτιθέμενες δηλαδή και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ανταποκριθούμε στο ύψος των προκλήσεων με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί θα πρέπει να αποστείλουμε στην Επιτροπή ένα ηχηρό μήνυμα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να καταβάλουμε μία προσπάθεια για να δείξουμε ακριβώς ότι φέρουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Αρχίζουμε με την τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές. Θα επαληθεύσουμε για την τροπολογία 17, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές μπορούν όλες οι ομάδες ε, να, ε, να, δείχνουν πολύ καλά, να ανεβάζουν καλά το χέρι ευκρινώς. Μπορούμε και πάλι. Τροπολογία 18. Υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, θα επαληθεύσουμε. Δεν ξέρω πολύ καλά. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίθηκε. 60 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 61 υπέρ, κατά. Θα επαληθεύσουμε για την 61 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Όχι. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. 22 υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε για την 22. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 24 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 62 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 62, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 25 υπέρ, κατά αποχές. Επαληθεύουμε για την 25. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε για την 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα επαληθεύσουμε. Σοσιαλιστές και ε, ΕΛΚ ψήφισαν υπέρ. Λοιπόν, 71 άρχεται η ψηφοφορία. 71. Τροπολογία 71. Ξαναρχίζουμε. Για την 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε για την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι πάντα η ίδια πλειοψηφία. πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Αν μπορείτε να μας... Δεν μπορώ να σας δω όλους καλά. 33 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε για την 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε για την 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ε, απαληθεύουμε για την 77, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ και κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε για την 79. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, άρχεται η ψηφοφορία για την 80, ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Επαληθεύουμε για την 82. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε για την 83 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές θα ε, ελέγξουμε για την 37. Ψήφισαν όλοι για την 37. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές 39 επαληθεύουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 40 υπέρ, ΕΛΚ, ΕΛΚ, 40 υπέρ, αποχές, 40, επαληθεύουμε, ψήφισαν όλοι, πέρα της ψηφοφορίας, εγκρίνεται, 41 υπέρ, κατά, αποχές, ας επαληθεύσουμε για την 41, Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 42 υπέρ και πάλι θα επαληθεύσουμε για τις 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για τη 43 Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Παραρτήματα 44 υπέρ κατά αποχές. σα ελέγξουμε για την 44. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 45 υπέρ. Θα ελέγξουμε για την 45. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Θα ελέγξουμε την 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε διαφορετικές πλειοψηφίες. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47. Θα ελέγξουμε για τη 47. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 48. Θα ελέγξουμε γιατί 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ψηφίστε τώρα. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 49. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για την 50 επίσης, άρχεται η ψηφοφορία. Είναι πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Τις σκέψεις 51 υπέρ, κατά, σοσιαλιστές πάλι. 51. Σοσιαλιστές ήταν κατά. Όχι, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία την πρώτη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε για την 53 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την τροπολογία 2 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 3 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε για την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά θα πρέπει να επαληθεύσουμε και για την πέντε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν βλέπω πολύ καλά ε, τα χέρια. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε για την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά δεν βλέπω πολύ καλά τα χέρια σας. 7. Θα ελέγξουμε για την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 54. Έχω ε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της 54, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Θα επαληθεύσουμε για την 9, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 55. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές. Θα επαληθεύσουμε για την 56. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές. Θα επαληθεύσουμε. 11 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, θα επαληθεύσουμε για τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλοι ψήφισαν πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13, 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε για την τροπολογία 15. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Φτάσαμε στο τέλος. Τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Έχουμε μικρή πλειοψηφία, εγκρίνεται όμως. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον εισηγητή. That και έτσι ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες και όποιος αποχωρεί να αποχωρεί ησύχως. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, περιμένουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής λόγω των απεργιών. Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Θα φτάσει όμως σε μερικά λεπτά. Θα υπενθυμίσω ότι έχουμε το επόμενο θέμα, πρόγραμμα δράσης για το φύλλο που έχουμε προσκεκλημένους από την Νιγηρία και το κοινοβούλιο τη, ξέρετε, στο κομμάτι που μοιραζόμαστε με την Επιτροπή των Γυναικών, με την κυρία Χάιτι Χάουταλα και πρόεδρο τη Επιτροπή των Γυναικών. Παρακαλώ να είσαστε όσο το δυνατόν πιο πολύ παρόντε. Έχουμε βουλευτέ γυναίκε τη ε, Νιγηρίας και νεαρές ε, γυναίκες από την Αφρική, η μία από τη Βραζιλία. Οι άλλοι περιμένουμε τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή, δεν ξέρω πόσο μακριά βρίσκεται και γιατί έχει πάρει αυτοκίνητο τέτοια μέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τώρα το 12 σημείο. Έχουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Πρέντα Παρόντα, για το θέμα της ρεύσης κατάστασης όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για την ε, πολιτική συνοχή, συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Έχουμε και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής θα μας εξηγήσει γιατί δεν υπάρχει έκθεση για το 2016 και το 2017. Είστε στη μετάβαση από ό,τι καταλαβαίνω για το 2030, αλλά οπωσδήποτε ο Γκάσπαρ θα μας εξηγήσει. Ο Γκάσπαρ Φροντίν εδώ. Τμήματάρχης της ΔΕΦΚΟ. Πολύ καλά τον γνωρίζουμε. Έχει ασχοληθεί με πολλά θέματα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ακούμε λοιπόν πρώτα την Επιτροπή και μετά στον μόνιμο συγητή μας, τον κύριο Πρέντα. Γκάσπαρ. Πήρες μια ανάσα. Ήταν κανθόδης ο δρόμος μέχρι να φτάσει εδώ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές. Κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ για αυτή την ανταλλαγή κάποιων ιδεών και πληροφοριών από την ε, πλευρά μας για την ε, συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος, όπως είπε και η Λίντα, πολύ σωστά. Από την προηγούμενη φορά που είχα έρθει να σας μιλήσω για τη συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Έχουν αλλάξει πολλά. Ήταν το 2015 τότε. Μεταξύ άλλαξε το θεματολόγιο και αρχίσαμε μέσα στο θεματολόγιο να υλοποιούμε τη συνοχή, προσπαθώντας να δούμε πώς μπορούμε να την ε, ενσωματώσουμε στο νέο θεματολόγιο και να πιέσουμε για την... Ε, και να βοηθήσει στην ε, ενίσχυση του επίπεδου υλοποίησης του νέου θεματολογίου, όπως ζητούσε άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο η Επιτροπή στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συνοχή, για την ΣΑΠ. Μας είχε ζητήσει το Συμβούλιο να ενσωματωθεί καλύτερα η ΣΑΠ στη νέα προσέγγιση για την υλοποίηση του θεματολογίου 2030 και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η καταγραφή ε, των εργασιών και των αποτελεσμάτων θα, να ενσωματώνει καλύτερα τα διδάγματα του παρελθόντος. Επίση το Κοινοβούλιο το 2014 μας είχε, το είχε πει μάλλον ότι η ΣΑΠ είναι κέριο στοιχείο για την υλοποίηση και την επιτεύξη της νέας, του νέου αναπτυξιακού θεματολογίου και μας είχε ζητήσει να αναλάβουμε ενεργό δράση εν προκειμένου. Δεν νομίζω να τη λοιπόν κανείς που όταν ε, συντάξαμε από κοινού το η νέα συνένεση για την ανάπτυξη ενσωματώσαμε σε αυτήν την ΣΑΠ, όπως άλλωστε και στο θεματολόγιο του 2030. Θα θυμάστε ότι αυτή η συνένεση, στην οποία συμφωνήσαμε τον Ιούνιο, πρώτον, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην ΣΑΠ, με σαφέστατους όρους πιστεύω, Δεύτερον, αναγνωρίζει ότι η ΣΑΠ είναι κέριο σημείο για την υλοποίηση του θεματολογίου του 2030, που όπως έχει ήδη υποθεί, χρειάζεται οπωσδήποτε και χρηματοδότηση, αλλά και πάνω απ' όλα ε, σαφή επιδίωξη των στόχων και των προτεραιοτήτων. Επίσης, ΑΠ πρέπει να καλύπτει όλα τα τμήματα και τους τομείς του θεματολογίου του 2030, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς όπως το εμπόριο, η οικονομία, το περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια των τροφίμων, μετανάστευση και ασφάλεια. Επίσης, η ιδέα για μία προσέγγιση από κάθε τομέα διακυβέρνησης έχει υπογραμμιστεί με ιδιαίτερη έμφαση. Και αυτό σημαίνει και για το μέλλον ιδιαίτερα ότι θα πρέπει και να γίνεται η εκ των προτέρων αξιολόγηση των συνεπειών των δράσεων μας, πριν αυτές αποφασιστούν δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα και η εκ των υστέρων αποτίμηση της εφαρμογής των αποφάσεων. Επομένως, πλέον έχουμε περάσει σε ένα νέο στάδιο, βγαίνουμε από τα τετριμένα και τη ρουτίνα στην υπόθεση ΣΑΠ, την βλέπουμε μέσα στο νέο θεματολόγιο 2030 και αυτή είναι η δουλειά όλων μας τον τελευταίο καιρό, μας απασχολεί πάρα πολύ. Η νέα δομή της Επιτροπής ε, που περιστρέφεται γύρω από έργα τα οποία διαχειρίζονται αντιπρόεδροι ε, μας βοηθεί περισσότερο να διαφυλάξουμε αυτή την έννοια της συνοχής για την, ανανεω... για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη επικεφαλής ε, μιας ομάδας έργου είναι ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς πρόκειται για την ομάδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη με συμμετοχή όλων των αρμοδίων επιτροπών και αντιπροέδρων και πρόκειται βέβαια για ένα πολιτικό όργανο μέσα από το οποίο εξασφαλίζεται η σε πολιτικό επίπεδο συνοχή. Σε ένα επίπεδο χαμηλότερο της ιεραρχίας, της υπηρεσίας, έχουμε μια διατομεακή ε, ομάδα, η υπηρεσιακή ομάδα για την αηφόρο ανάπτυξη που οργανώνει ο Γενικός Γραμματέας αλλά ταυτόχρονα συμμετέχουμε όλοι από διάφορες ε, γενικές διευθύνσεις. Πρόκειται για μια ομάδα στην οποία θα συναντηθεί το έργο της ΣΑΠ με το, με λοιπό και όλο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ανάπτυξη. Και παράλληλα αυτή η ομάδα θα αναθεωρεί ε, περιοδικά την πρόοδο, θα αξιολογεί την πρόοδο στην ΣΑΠ. Δηλαδή θα έχουμε και εσωτερική αλλά και εξωτερική πτυχή στο έργο αυτό της αξιολόγησης που πιστεύουμε ότι θα μας οδηγήσει σε μια πλήρως ενσωματωμένη στο όλο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνοχή για την, της αναπτυξιακής πολιτικής. Για να ενισχυθεί περαιτέρω ο μηχανισμός ε, που έχουμε από το παρελθόν, ε, στο παρελθόν ήδη καθιδρύσει, έχουμε αξιοποιήσει την αναθεώρηση, το, εργα, εργαλείο, την εργολιοθήκη μάλλον, της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών σε μια αξιολόγηση, μια σε στάδιο της ΣΑΠ. Και έτσι ο όρος αντίκτυπος στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει εγγεγραμμένο σε όρους ρητούς, ενώ πριν γινόταν λόγος μόνο για αντίκτυπο σε τρίτες χώρες. Τώρα μιλούμε για αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό το εργαλείο κάθεται στρατηγική σημασία για την αξιολόγηση του αντικτύπου των διαφόρων αποφάσεων της Επιτροπής αλλά της, Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι όρος ενσωμάτωσης της ΣΑΠ και ταυτόχρονα έχουμε και την ενσωμάτωση του έργου της ΣΑΠ διαρθρωτικά, δομικά, στο όλο έργο της Επιτροπής. Πράγμα το οποίο, αν δεν με συχνά έχει στήσει το κοινοβουλίο σας να μην ε, μπαίνει στην γωνία η να, να μην βρίσκεται σε μια γωνία ΙΣΑΠ, αλλά να ενσωματώνεται ως κανονικός, ως φυσιολογικός όρος ε, σε όλο το έργο της Επιτροπής. Και επίσης έχουμε το ε, Συμβούλιο Ρυθμιστικής Επαλήθευσης, το Regulatory Scrutiny Board, το οποίο έχει βέβαια ως ρόλο την αξιολόγηση των νομοθετικών παρεμβάσεων και με ιδιαίτερη έμφαση τώρα ε, στο ε, έργο το σχετικό με τη ΣΑΠ, το οποίο έχει ενσωματωθεί στα καθήκοντά του και ελπίζουμε ότι θα μας υποστηρίξει εν προκειμένου. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να ενσωματώνουμε την ΣΑΠ στις νέες δομές ε, εργασίας, συνεργασίας εν ώψη του θεματολογίου του 2030 με ανάπτυξη των εσωτερικών όσο και εξωτερικών πτυχών της πολιτικής μας για, την, ε, για τις εκθέσεις καταγραφή αποτελεσμάτων. Θέλω να σας επισημάνω το εξής. Πρώτον, όπως γνωρίζετε ίσως, στις 20 Ιουνίου του 17 με τα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει την πρώτη ιστορική αναθεώρηση έκθεση για την υλοποίηση του θεματολογίου 2030 εν ώψη της υποβολής ε, στην ε, Σύνοδο το 2019 στην Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου. Ξέρετε ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη που, που ανακοινώνει δέσμευση για μια κοινή έκθεση από τα κράτη-μέλη για τις προσπάθειες ε, για την υλοποίηση του θεματολογίου και βέβαια παρουσίασε το 2019 στην Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου, στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου. Ε, και πρέπει να κοιτάξουμε με ιδιαίτερη έμφαση την βελτίωση της έκθεσης πεπραγμένων Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξέταση μιας σειράς από επιλογές για μια ε, ολοκληρωμένη υποβολή ε, έκθεση πεπραγμένων, που θα λαμβάνει υπόψη δηλαδή όλα τα ανωτέρω. Και εδώ ιδιαίτερα κοιτάμε πώς μπορούμε στο μέλλον η ε, έκθεση πεπραγμένων ΣΑΠ θα μπορούσε να ενταχθεί στην συνολική έκθεση πεπραγμένων. Ως στοιχείο κέριο των συνολικών προσπαθειών μας για την υλοποίηση του θεματολογίου 2030. Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες ε, σχετικές με την βελτίωση της ε, υποβολής εκθέσεων. Πρώτα απ' όλα, υποβολή εκθέσεων για την υλοποίηση της, από τις αντιπροσωπείες, με πολύ, σημαντικό, βέβαια, πολύ σημαντική διάσταση εδώ, διότι οι αντιπροσωπείες είναι αυτές οι οποίες έχουν την καλύτερη δυνατότητα να δουν ε, τι είδους αντίκτυπο μπορεί να φέρει η ΣΑΠ στις ε, επιμέρους χώρες. Αυτές μπορούν να κάνουν την, ε, τον απολογισμό. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε λοιπόν αυτόν τον απολογισμό, τον καθιστούμε ετήσιο, ετήσιο λοιπόν απολογισμό από τι αντιπροσωπείες. Επίσης τον επεκτείνουμε σε όλες τις αντιπροσωπείες. Το 2016 νομίζω ήταν 84 ε, οι αντιπροσωπείες που υπέβαλαν απολογισμό καλύπτοντας 110 διαφορετικές χώρες με τεράστια βέβαια αύξηση σχέση με το προηγούμενο έτος και ταυτόχρονα σχεδόν ε, κάλυψη όλης της υφηλίου. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί αλλά πλησιάζουμε. Δεν θα μπω στις ε, λεπτομέρειες των, ε, ε, της ανταπόκρισης και των ε, τομέων που καλύφθηκαν, αλλά πάντως έχουμε με κύριο άξονα το εμπόριο, πολύ θετικό αντίκτυπο και απολογισμό του εμπορίου, του εξωτερικού εμπορίου και του αντίκτυπου του στις χώρες. πολλά σχόλια σχετικά με την αλία και μάλιστα την παράνομη, αλία, πολλές ανησυχίες. Και βέβαια πολλά, πολλά, πολλά σχόλια στις εκθέσεις αυτές αναφέρονται στην μετανάστευση. Σε σχέση με αυτά που κάνουμε λοιπόν για τον απολογισμό και τη ΣΑΠ και την προσπάθεια να αξιολογήσουμε τις προσπάθειές μας στη ΣΑΠ, όπως θα ξέρετε ίσως έχουμε ξεκινήσει μια εξωτερική αξιολόγηση της ΣΑΠ, όπως έχει ζητήσει τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο, ένα έργο ογκώδες με αξιολόγηση των στόχων και τις υλοποίησης τους στις επιμέρους περιοχές ως προς την αναίφορο ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας. Τι έχει φέρει η ΣΑΠ. Η αξιολόγηση δηλαδή προσπαθεί να καλύψει τρία επίπεδα. Εξωτερική αξιολόγηση. Κοιτάει καταρχάς εάν τα εργαλεία τα οποία έχουμε προβλέψει αξιολόγηση αντικτύπου, αξιολόγηση περιεχομένου, εμ, κύκλος κατάρτισης φέρνουν αποτελέσματα. Δεύτερον, εξετάζει αν τα συγκεκριμένα εργαλεία έχουν αντίκτυπο ως προς τις διάφορες περιοχές ε, εμπόριο, γεωργία λοιπά που έχουμε ε, επιλέξει. Δηλαδή αν, αλλάζουν αυτές οι πολιτικές χάρη στα εργαλεία της ΣΑΠ και τρίτον, εάν αυτές οι αλλαγές πολιτικής όταν υπάρχουν έχουν θετική θετικό αντίκτυπο στις χώρες αυτές, ε, χώρες εταίρους για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, ή φορονάπτυξη. Και επίσης Έχουμε μια σειρά από ερωτήσεις, από στήλη, ερωτηματολόγια από πλευρά της Επιτροπής Δεύτερες Χώρες, από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Βοήθειας, ε, με απαντήσεις που στέλνονται προς μια κεντρική μονάδα και μετά βεβαίως θα γίνουν και οι αυτοψίες για να δούμε αν ε, οι εκθέσεις έχουν ε, σχέση με την πραγματικότητα, εκθέσεις οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στο πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ παράλληλα γίνεται μια ευρεία διαβούλευση επί 12 εβδομάδες με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να συλλεγούν οι απόψεις και οι ιδέες τους ή τα σχόλιά τους για κάθε τομέα και από εκεί θα προκύψει η αξιολόγηση. Όπως είπα θα πρόκειται και μια ανεξάρτητη αξιολόγηση, δεν ελέγχουμε εμείς την αξιολόγηση αυτή της ΣΑΠ, την εξωτερική, αλλά βάσει αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή θα αντλήσει συμπεράσματα, ενδεχομένω δε και να δώσει απαντήσει σε κάποια από τα σχόλια της αξιολόγησης σε ένα έγγραφο εργασίας εσωτερικό, staff working document, που θα υιοθετηθεί μέχρι τα μέσα του 2018. Άρα θα έχει και συνέχεια αυτή η εξωτερική αξιολόγηση. Αυτά λίγο πολύ. Όσα κάνουμε για την προσαρμογή της ΣΑΠ στο θεματολόγιο 2030. Μας απασχολεί αρκετά, όπως βλέπετε, είναι, μας δίνει αρκετή δουλειά. Είναι πολλά θέματα που μας απασχολούν. Ταυτόχρονα για να κλείσω έχουμε ε, ε, περιλάβει ένα εργαλείο ηλεκτρονικής ε, μάθησης e-, e-learning tool ε, στην SAP. Αυτό αφορά το προσωπικό μας αλλά και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί τι είναι SAP, τι εργαλεία έχει, τι μπορεί να κάνει. Είναι ενδιαφέρον πιστεύω. Ενημερωτικό εργαλείο για όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με τη ΣΑΠ. Αυτά από μένα προς το παρόν και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να δώσω απαντήσεις ή σχόλια σε οποιοδήποτε θα μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα διότι η έκθεση αυτή αυτή θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για να την αποτιμήσουμε. Έχουμε όμως και τον εισηγητή μας, τον κύριο Κριστιαν Πρέντα, ο οποίος θα κάνει μία εισήγηση. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. πρότεινα αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή έτσι ώστε να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις της ΣΑΠ και της ε, διάδρασης με την ατζέντα του 2030. Αυτά τα ε, μέτρα που προτείνεται με ικανοποιούν, ο τρόπος δράσης δηλαδή. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ορισμένα σημεία υποβάλλοντας και ορισμένες ερωτήσεις. Προς την Επιτροπή είπατε ότι η ΣΑΠ είναι ένα κομβικό στοιχείο για την εφαρμογή της Ατζέντα 2030 και των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συλλογιστούμε για να δούμε πώς η ΣΑΠ θα ε, εμπλακεί στην Ατζέντα 2030. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει στη δράση ε, έτσι ώστε να προωθήσουμε και την ε, συνεκτική πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο, στο ίδιο μήκος κύματος με όλους τους διεθνείς εταίρους και ιδιαίτερα τα Ηνωμένα Έθνη και φαίνεται ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα, όχι δηλαδή μέσα σε μία δεκαετία. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι η διετής έκθεση είναι ο βασικός μηχανισμός που επιτρέπει στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν για τη ΣΑΠ. Δεχτήκαμε την ιδέα ότι η έκθεση αυτή υποβάλλει τα βασικά ε, αιτήματα, αλλά ε, δεν ε, λάβαμε υπόψη την ε, μέγιστη δυνατή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς μπορείτε, πώς σκέφτεστε να διατηρήσετε αυτό το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια είναι ένας βασικός φορέας της ΑΠ στην έκθεσή μου κίνησα την ιδέα η οποία υποστηρίχθηκε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη ΣΑΠ για να δούμε πώς θα λειτουργήσει έμπρακτα η ΣΑΠ και ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός σε αυτό το πλαίσιο. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στην πρόοδο της ΣΑΠ θα πρέπει να συζητηθεί στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο. Αυτό το είπα κατά τις ανταλλαγές μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκέφτεστε από αυτού. Δηλαδή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ΣΑΠ, συνάντηση υψηλού επίπεδου. Τέλος, ε, αναφερθήκατε σε αυτήν την ομάδα επιτρόπων που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα ως προς τη ΣΑΠ και την Ατζέντα 2030. Γιατί μιλήσαμε για συνεδριάσεις, τις οποίες προείσταται ο Επίτροπος Τίμερμανς και θα ήθελα να μου πείτε μέχρι του χρόνου τι βλέπετε να δρομολογείτε. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα ως προς τις ε, σχέσεις μεταξύ των διαφόρων αντιπροσωπιών. Υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των αντιπροσωπιών και αυτό το χαιρετίζουμε από πλευράς Κοινοβουλίου δεν έχουμε πολλές πολιτικές ομάδες εδώ, δυστυχώς, που να παρίστανται. Έχουμε μερικές βέβαια, αλλά ελπίζω να συμφωνήσουν μαζί μου για να χαιρετήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κριστιαν Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα χρειάζεται τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. των εκθέσεων βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την συνοχή στην πολιτική μας για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, που είναι στην προτεραιότητα. Χρειάζεται λοιπόν η συνοχή στους διάφορους τομείς ε, της πολιτικής ε, όπως, το όπως η γεωργία, η ενέργεια, η πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας και οτιδήποτε άλλο πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα το στόχο αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη κάποια πρόταση ή κάποια αποτελέσματα ή συμπεράσματα που μπορείτε να διτυπώσετε σε σχέση με την έκθεση για το πρώτο κομμάτι ως το 2018, για το πρώτο τρίμηνο του 2018, εάν δηλαδή τα κράτη-μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πράγματι ενσωματώσει την συνοχή αυτή, την ε, υποχρέωσή τους για μια συνεκτική πολιτική και αν την έχουν αναλάβει ως υποχρέωση. ώστε να εκφράζεται σε όλους τους τομείς της πολιτικής. Ε, με αισθάνομαι μια κάποια απογοήτευση που δεν έχουμε ε, που δεν έχουμε λάβει έκθεση, που δεν θα έχουμε φέτος έκθεση, αλλά ελπίζω του χρόνου να είναι καλύτερη, πληρέστερη, όπως μας υποσχεθήκατε. Όλα αυτά ωραία ακούγονται. Μέχρι όμως να έρθει αυτή η νέα μορφή έκθεση. δεν θα έχουμε καμία έκθεση. Και απολογισμό για την αναπτυξιακή βοήθεια. Επομένως, τι γίνεται μέχρι να υπάρξει αυτή η νέα εκδοχή, η νέα μορφή εκθέσεων και να λειτουργήσει, γιατί δεν συνεχίζετε την παλιά μορφή που είχαμε τόσο καιρό. Έτσι ώστε και εμείς να είμαστε ενήμεροι. Είναι θλιβερό το ότι δεν έχουμε έκθεση για την ΣΑΠ φέτος. Και το θεωρώ σοβαρό έλλειμμα. Είπατε και εσείς κύριε Πρέντα άλλωστε ότι δεν βλέπετε αρκετά σαφή ή επαρκή την συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαδικασίες αυτές. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει και εμείς από πλευράς μας να ενεργοποιηθούμε, να δραστηριοποιηθούμε και να πούμε τι ακριβώς θέλουμε. Ο κύριος Γκερέρος παραδείγμα παραδείγματι, ο συντονιστής και μόνιμος εισηγητή στην ανθρωπιστική βοήθεια πολύ συχνά στις συνεδριάσεις των συντονιστών μας δίνει τις ιδέες του για το τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα έπρεπε να κάνουμε και ίσως και για τη ΣΑΠ θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε αντίστοιχες προτάσεις για περισσότερη κινητικότητα. ώστε να μπορούμε και στο μέλλον να παρακολουθούμε καλύτερα αυτές τις εκθέσεις και να συμμετέχουμε σε αυτές. Ευχαριστώ κύριο Σκοράου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπη για την παρουσίαση και συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έγιναν από την αδελφό Μαρία. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω στην βασική αρχή της ΣΑΠΑ οι πολιτικές των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται στην συνεκτικότητα των πολιτικών των αναπτυξιακών. Αλλά δεν βλέπω πολύ συνεκτικότητα ε, με τον τρόπο της κατανομής των πόρων. Η περισσότερη υποστήριξη χρηματοδοτική βασίζεται στις πολιτικές μετανάστευσης που δεν έχουν καλή παρακολούθηση και έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση προόδου στα πλαίσια της ΣΑΠ. Νομίζω ότι ε, επίση στις συμφωνίες δεν έχουμε συνεκτικότητα. Θα πρέπει στις συμφωνίες να βρούμε έναν τρόπο ελέγχου για να δούμε, για να υπάρξουν ε, μειώσεις του αριθμού των μεταναστών. Νομίζω ότι έχουμε 3 δισεκατομμύρια τα δύο έτη και άλλα 3 δισεκατομμύρια αφού αυτά τα χρήματα χρησιμοποιηθούν πλήρως στο τέλος, μέχρι το τέλος του 2018. Υπάρχει λοιπόν χρηματοδότηση χωρίς συνεκτικότητα, ε, διότι η χρηματοδότηση δίνεται σε χώρες όπως η Τουρκία, όπου δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν έχουμε κριτήρια για να εγγυηθούμε ε, την, ε, τα αποτελέσματα για να δούμε αν οι πόροι κατανέμονται και διοχετεύονται και χρησιμοποιούνται σωστά. Χρειάζομαι και χρειαζόμαστε ένα σύστημα παρακολούθησης για να έχουμε μια αναλογία ανάμεσα στα χρήματα που ξοδεύονται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα προσθέσω και τον εαυτό μου στον κατάλογο. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε συγητής Διαρωτώ με, η Μαρία μίλησε για το πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ίσως θα πρέπει να επιλέξουμε ορισμένα σημαντικά θέματα για τη ΣΑΠ. Βεβαίως, καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι αν έχουμε έκθεση κάθε δύο χρόνια, ίσως ε, υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ίσως δεν βλέπουμε τα πράγματα εις βάθος. Ίσως ε, θα χρειάζεται πιο πολύ εις βάθος εξέταση των διαφόρων θεμάτων, αλλά ίσως θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους τομείς που μας απασχολούν περισσότερο και να δούμε τις λεπτομέρειες αυτών των τομέων. Ίσως αγροτική πολιτική, αλλιευτική πολιτική, θα μπορούσε να είναι η ενεργειακή πολιτική, η εμπορική πολιτική, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάτι το ειδικό μέσα σε κάθε τομέα. Ίσως ε, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος ε, να διεκπαιρεώσουμε τη συζήτηση καλύτερα. Και πάλι στον Κάσπαρη ερώτησή μου, όταν κάνετε αυτήν την έρευνα με την υπηρεσία σου, ε, πώς βεβαιώνεστε για την άσκηση. Βεβαίως, πώς ε, έχετε τα αιτήματα από πολιτικούς, τα έντυπα, ε, παρακολουθήστε ε, τα, το, τα θέμα του φύλου, το θέμα του περιβάλλοντος και το ελέγχετε και το πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε πραγματικά θέματα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τα συγκεκριμένα αυτά θέματα και όχι να έχουμε γενικότητες στα, στις, όπως είναι στις δεκθέσεις των μεγάλων διοίκησεων. Κανείς δεν ζήτησε τον λόγο. Ξαναδίνω λοιπόν πάλι τον λόγο στον Κάσπαρ. Πολύ ενδιαφέρουσες και από της είναι οι ερωτήσεις και θα σας δώσω, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Καταρχήν θα πρέπει να γίνει μία προσαρμογή ε, της ΑΠ στην ατζέντα του 2030 και αυτό αποτελεί μία πολύ μεγάλη ευκαιρία ε, έτσι ώστε να μην συμπληρώνουμε τα τετραγωνίδια απλώς, αλλά να κάνουμε μία δουλειά επί της ουσίας. Εργαζόμαστε επ' αυτού. Μιλήσατε για την βιώσιμη ανάπτυξη και υπάρχει ε, μία σύγχυση ως προς την ε, πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής για την βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν η ατζέντα του 2030 αναφέρεται στην ε, συνεκτική βιώσιμη ανάπτυξη, αφορά την συνοχή που χρειάζεται ολοκληρωτικά για να εφαρμοστεί η ατζέντα, δηλαδή η συνοχή όλων των πολιτικών, ανθρώπινα δικαιώματα, χρηστή διακυβέρνηση, κλιματικές αλλαγές και ούτω καθεξής. Τώρα, η ΣΑΠ, όπως αναφέρεται στις συνθήκες, είναι πιο Εστιασμένοι, δηλαδή για την ΣΑΠ, οι συνθήκες μας ζητούν να ελέγξουμε το κατά πόσο οι δράσεις μας σε άλλες πολιτικές έχουν επιπτώσει στις αναπτυσσόμενες χώρες και να αποτιμήσουμε αυτή την επίπτωση. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο θεωρούμε ότι υπ' αυτή την έννοια η ΣΑΠ θα ήταν ένα χρήσιμο μέσο για να εργαστούμε για μια καλύτερη πολιτική συνοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε μέσα ε, και εδώ υπάρχουν και οι δεσμεύσεις της συνθήκης, των συνθήκων που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ας χρησιμοποιούμε λοιπόν, ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα ως οικοδομικά υλικά για να χτίσουμε την πολιτική μας μέσα στα πλαίσια της συνοχής ε, για την ατζέντα του 2030. Και αυτό είναι το φιλοσοφικό μας υπόβαθρο, αυτή είναι η συλλογιστική μας, γιατί πολλές φορές σε αυτές τις συζητήσεις καθώς και σε άλλες Λέγατε στην Επιτροπή ότι αυτό που κάνουμε για τη ΣΑΠ είναι πολύ καλό, αλλά υπάρχουν περιορισμένες επιπτώσεις. Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι έχετε μερικός δίκιο, αλλά τώρα υπάρχει μία ατζέντα εσωτερική και εξωτερική. Θα συζητήσουμε πολιτικές και εδώ θα μιλήσουμε και για τις ε, εξωτερικές επιπτώσεις όλων των πολιτικών και εδώ εντάσσεται και η ΣΑΠ. Και αυτό θα οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα και ακριβώς αυτό επιθυμούμε, δηλαδή να εντάξουμε τη ΣΑΠ στην Ατζέντα 2030. έτσι ώστε να έχουμε ένα διπλό εγχείρημα με ένα απότερο στόχο. Αυτή είναι η συλλογιστική μας. Ε, θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί μας και να λογοδοτούμε σε εσά γιατί το Κοινοβούλιο μας βοηθά ιδιαίτερα για την οικοδόμηση της ΣΑΠ και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε σε όποιο τομέα το επιθυμείτε. Τώρα, ως προς την εξειδικεμένη εξειδικευμένη πρόταση ενός Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου για τη ΣΑΠ, ε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Αλλά θα πρέπει η ΣΑΠ να συνδεθεί με την Ατζέντα 2030 για να μπορεί να γίνει μια συζήτηση υψηλού επίπεδου. Ως προς το γεγονός ότι χρειάζεται συνοχή για όλες τις πολιτικές, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε επακριβώς, αλλά να το συνδέσουμε με την όλη εργασία της Επιτροπής για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ως προς την αξιολόγηση, την έκθεση αξιολόγησης που θα λάβετε το 2018, δεν έχουμε ακόμα δεδομένα γιατί πρόκειται για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Όταν ολοκληρωθεί θα δούμε ποια είναι τα ευρήματα και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα. Δηλαδή, έχετε μία ανεξάρτητη αξιολόγηση και την αποτίμηση της Επιτροπής του Χρόνου. Έτσι, θα μπορέσουμε να λογοδοτήσουμε, να αποτιμήσουμε την κατάσταση και αυτό σε σχέση με την Ατζέντα 2030. Και γι' αυτό νομίζω ότι εντάσσεται πολύ καλά στο ολοεγχείρημα της Ατζέντα 2030. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη έκθεση για την Ατζέντα 2030. Ως προς το πρότυπο συνοχής, ένα ζήτημα και μόνο. Ναι. Σε σχέση με τη συμφωνία με την Τουρκία, η ΣΑΠ δεν λέει ότι ο αναπτυξιακός στόχος θα πρέπει να υπερισχύσει σε άλλων ε, θεμητών στόχων ή στόχων νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, όταν λαμβάνετε αποφάσεις σε άλλους τομείς θα πρέπει να αποτιμήσετε τις επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν θετικές συνέργειες ή, εν πάση να απαλύνουμε τα αρνητικά. Ως προς το τελευταίο ερώτημα, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε πιο εξειδικευμένοι για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη επίπτωση φυσικά. Υπάρχουν δύο τρόποι, δηλαδή η μεθοδολογία, τα μέσα, η εργαλειοθήκη, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια αυτής της πορείας και αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε, αυτά θα πρέπει να τα συνδέσουμε με την καθημερινή εργασία της Κομισιόν. Μετά όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους τομείς που θα δράσουμε. Έτσι ώστε να δούμε πού μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας και πού μπορούμε να διαδράσουμε και να έχουμε επιπτώσεις γιατί φυσικά οι αλλαγές θα επέλθουν σε συγκεκριμένους τομείς. Και σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να δούμε τα πράγματα. Αυτά μπορώ να σας πω σε αυτό το στάδιο των εργασιών. Ο κύριος Πρέντα, Κριστιαν, θέλεις να σχολιάσεις? Όχι. Όχι, όχι, σε αυτό το στάδιο όχι. Να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κύριο Φροντίνη Όπως ξέρετε, πρόκειται για μια διαδικασία ολοκλήρησης και μια εμβάθυνση και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να επιλέξουμε ένα-δύο θέματα πριν από το τέλος της θητείας, γιατί ο χρόνος ε, περνάει. Είμαστε ήδη, φτάσαμε στο Σεπτέμβριο 2017, γι' αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε ένα ε, τομέα που θα μας απασχολήσει εις βάθος μετά τα Χριστούγεννα. Και μετά θα έχουμε και αυτή την έκθεση, γιατί πιστεύω θα την έχουν την έκθεση το καλοκαίρι του 2018. Τη δική σας έκθεση, δηλαδή την, την ανάλυση του ανεξάρτητου φορέα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι και μετά, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε λίγο νωρίτερα, να επιλέξουμε ορισμένους τομείς για να δούμε ποιοι είναι οι πιο δύσβατοι τομείς για τη ΣΑΠ για να δούμε και την κλίμακα του ζητήματος. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Φροντίνη από την Κομισιόν. Τώρα έχουμε μία κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΦΑΜ σε 10 λεπτά. Βλέπω ότι η υπεύθυνη έρχεται τώρα. Θα σταματήσουμε και έχουμε και ε, ειδικούς επισκέπτες και θα ήθελα να πω ότι σήμερα το απόγευμα αρχίζουμε στις 2.30, όχι 3, 2.30, όχι 3. Και αυτό γιατί τελειώνουμε νωρίτερα για να ψηφίσουμε για το βραβείο Ζαχάροφ στις 5 μαζί με την ΑΦΕΤ. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε σε 10 λεπτά.